Pan Przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ε, συνεδρίασής μας είναι η έκθεση του κυρίου Σαλβατόρ Γκαρίκα Πολέντο σχετικά με την επένδυση στο μέλλον. Είναι ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμού. Το λόγο θα πάρει καταρχήν ο ίδιος ο εισηγητής. Κύριε Σαλβαδόρ Γκαρίγα Πολέντο έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επιτρόπε Λεβαντόφσκι, συνάδελφοι, εδώ και 23 χρόνια εκδίδουμε δημοσιονομικέ προοπτικές σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους.